Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε προσκεκλημένοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής για σήμερα. Έχετε το σχέδιο εμερήσιας διάταξης. Μπορούμε να το εγκρίνουμε. Έχετε προτάσεις τροποποίησης, όχι. Θεωρείται λοιπόν η εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη ως έχει. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της 3ης Δεκεμβρίου 2014. Προτείνω όσοι ήθιστε, αν δεν ε, γύρει κανείς καμία αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Ωραία. Τρίτον, πάρα πολύ σύντομες ανακοινώσεις της Προέδρου. Άρχισε η νέα κοινοβουλευτική χρονιά για την Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας πω ότι θα παραθέσουμε δεξίωση για όλα τα μέλη, τακτικά, αναπληρωματικά, προσκεκλημένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Λετωνική Προεδρία ε, και τους βοηθούς και συνεργάτες εδώ Εκτό τη αιθούση, απόψη μετά τη λέξη συνεδρία στις 6.30. Εύκολα το βρείτε. Υπάρχει ένα χώρο εδώ. Αυτή ήταν η ε, σύντομη ανακοίνωση που είχα να σα κάνω. Και θα περάσουμε στο πρώτο ουσιαστικό θέμα για σήμερα. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να καλωσορίσουμε την πρώην συνάδελφό μας. Την κυρία Κορίνα Κρέτσου, την καλωσορίζουμε και πάλι στην Επιτροπή μας υπό τη νέα της ιδιότητα ε, ως αρμόδια επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Στο μέλλον πολιτική συνοχή θέλουμε να εστιαστεί σε δύο θέματα, να κλείσουν τα προγράμματα της προηγούμενης περίοδου 2007-2013, να δούμε τι αντίκτυπο είχαν και για ποιο λόγο δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια όλα. Και το δεύτερο είναι η κατάσταση ε, των πραγμάτων μετά την έγκριση των προγραμμάτων 2014-2020 καθώς αρχίζει η υλοποίηση και εφαρμογή τους. Ήδη από τώρα μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες βασικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα έτη. Να ενισχύσουμε και την αστική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής, μια προσέγγιση με βάση ε, τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις, μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές ενδιάμεσα αναθεώρηση του πολίτου του μεσονομικού πλαισίου. Η συσχέτιση των στρατηγικών επενδύσεων με τα σημερινά ταμεία, τα επιδυτικά και τα διαρθωτικά. Έχουμε λοιπόν μια σειρά θεμάτων να συζητήσουμε με την Επίτροπο, όχι μόνο σήμερα και στο μέλλον. Θα ακολουθήσουμε τη συνήθη διαδικασία. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Επίτροπο για να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή και στη συνέχεια στα μέλη για να κάνετε ερωτήσεις. Αρχίζοντας βέβαια από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων σε ένα πρώτο γύρο. Αν συμφωνείτε μπορούμε να συνεχίσουμε και να δώσουμε αμέσως το λόγο στην Επίτροπο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα ολόθερμα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να επιστρέψω στην Επιτροπή σας μετά από την ακρόαση του Σεπτεμβρίου. Και ξέρετε ότι πάντα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα παρευρίσκομαι εδώ πέρα σε εργασίες της Επιτροπής σας, διότι ε, νομίζω ότι από κοινού μπορούμε και μόνο από κοινού μπορούμε να σημειώσουμε επιτυχία και πρόοδο στον τομέα τη περιφερειακή πολιτική. Λοιπόν, καταρχά εύχομαι καλή χρονιά, ολογία και ευτυχία και πολλέ επιτυχίε για εσά και τι οικογένειέ σα. Όπω σα είπα, πέρασαν τέσσερι μήνε από την ακρόαση του Σεπτεμβρίου, μία σύντομη περίοδο για μένα και ξέρω βέβαια ότι κι εσείς την περίοδο αυτή αρχίσατε να επεξεργάζεστε διάφορες ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, αντιμετωπίζοντας διάφορα σημαντικά ζητήματα για την περιφερειακή πολιτική. Και προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική καρποφόρα συζήτηση μαζί σας για τις εκθέσεις αυτές. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τέσσερις αυτοί μήνες ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι και με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να σα παρουσιάσω τα πρώτα αποτελέσματα τη δράση μα σε τρει βασικού τομεί. Πρώτον, η έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων, η εφαρμογή των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 και επίσης συμβολή της πολιτικής συνοχής όσον αφορά το σχέδιο επενδύσεων και την δέσμη μέτρων του Προέδρου Γιούνκερ. Όσον αφορά την έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ανησυχίε που είχατε εκφράσει τον Νοέμβριο στο ψήφισμά σα, όπου είχατε πει ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνδυνο να υπάρχει καθυστέρηση στι πληρωμέ και κατά αυτόν τον τρόπο να μην μπορούν οι εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ να χρησιμοποιήσουν εγκαίρω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδίω σε μια περίοδο κρίση. Και εμά λοιπόν μα ανησυχεί αυτό και ξέρουμε ότι πάρα πολλέ περιφέρειε στην Ευρώπη ήδη υποφέρουν πάρα πολύ τα τελευταία 7 χρόνια εξαιτία οικονομική κρίση που πλήττει την Ήπειρό μα. Και θεωρούμε ότι μπορούμε στα πλαίσια τη πολιτική περιφερειακή πολιτική, στα πλαίσια τη περιφερειακή πολιτική, να δώσουμε περισσότερα κονδύλια προ τι περιφέρειε αυτέ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει την εργασία τους, δεν θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να περιμένουν ακόμα περισσότερο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουμε ήδη κάποια από τα αποτελέσματα. Το Δεκέμβριο εγκρίναμε 158 επιχειρησιακά προγράμματα με δύο σημαντικά ταμεία, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης έχουμε πλέον 40 επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα ακολουθήσουν στο μέλλον στα πλαίσια της διαδικασίας μετακύλησης, μεταφοράς των προγραμμάτων αυτών στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Γενικά αυτά αντιστοιχούν στο 75% όλων των προγραμμάτων όσον αφορά το στόχο για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τους τελευταίους 12 μήνες ένα 63% των προγραμμάτων του στόχου ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης έχουν εγκριθεί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόνο 15% το 2007, δηλαδή το πρώτο έτος της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πάει πολύ καλά αυτή τη φορά. Ακούσαμε επίση τι ανησυχίε σα τον Οκτώβριο του 2014 και είχατε πει τότε ότι είχατε καταβάλει πάρα πολύ σημαντικέ προσπάθειε, ιδίω στου τελευταίου μήνε Τη προγραμματικής περίοδου που έλεγε το 2014 για να εγκριθούν ακόμα περισσότερα προγράμματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε εγκρίνει ακόμα περισσότερα προγράμματα, είχε ασκηθεί πίεση επίση από τα κράτη-μέλη. Ξέρετε όμως ότι ήδη από τότε είχα πει ότι σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να κάνουμε συμβασμούς όσον αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων, ότι δεν θα έπρεπε να βιαστούμε πάρα πολύ διότι τα επιχειρησιακά αυτά προγράμματα τα οποία εγκρίνουμε αυτή την περίοδο αποτελούν το γενικότερο πλαίσιο δράσης για τα επόμενα 10 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά και πολύ προσεκτικά. Γνωρίζω βέβαια ότι επί τόπου υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που χρειάζονται τη χρηματοδότηση αυτή, αλλά δεν μπορεί αυτή να επέλθει με έναν οποιοδήποτε τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι η πολιτική αυτή δεν είναι απλή μεταφορά χρημάτων, δεν είναι μια φιλανθρωπική πολιτική, αλλά είναι μια σοβαρή περιφερειακή πολιτική, η οποία ενέχει τόσο υποχρεώσει όσο και δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν του επόμενου έξι μήνε θα προσπαθήσει να εγκρίνει τα πιο ποιοτικά προγράμματα και κατά αυτόν τον τρόπο θα δείξει την πιο υπεύθυνη στάση την οποία μπορεί να δείξει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε διάφορε συγκεκριμένε διαδικασίε και να καταφέρουμε να εντάξουμε εκ νέου στον προπολογισμό τα ποσά εκείνα τα οποία δεν είχαν καταβληθεί κατά το 2014. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μια αναθεώρηση και του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο θα εγκρίνουμε μια τέτοια τροποποιητική πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και θα γίνει αυτό βέβαια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη Λετωνική Προεδρία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τελικά μία επικοδομητική αναθεώρηση του προγράμματος αυτού, προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε και όλα τα εκκρεμή προγράμματα τη περιφερειακή πολιτική. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα αυτό, είμαι πεπισμένη ότι τα εκκρεμή προγράμματα θα μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε μέχρι τον Μάιο του 2015. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα αυτό, αλλά εξαρτάται και από την πολιτική βούληση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των προγραμμάτων 2007-2013, έχει σημειωθεί πρόοδος στην χρήση των ταμείων αυτών για την περίοδο αυτή. Τα πράγματα είναι αρκετά θαρρυντικά. Η χρησιμοποίηση των ταμείων πέρασε από το 59% της κατανομής χρηματοδότησης στα τέλη του 2013 στο 75% για τα τέλη του 2014. Με άλλα λόγια λοιπόν, 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε απαιτήσει πληρωμών καταβλήθηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες του 2014. Δυστυχώς όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές δυσκολίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση αυτή. Και ως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής έχω έρθει ήδη σε επαφή με τα κράτη-μέλη αυτά που έχουν ε, χαμηλά ποσοστά απορρόφησης και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μια ειδική task force για την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων προκειμένου να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σίγουρα το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο και εγώ θα ταξιδέψω προφανώς στις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα έρθω σε επαφή με τέρους, με εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών, προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους ε, δικαιούχους τους. Ξέρετε όμως ότι στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής μιλάμε για κοινή διαχείριση και κοινή ευθύνη. Οποιαδήποτε προσπάθεια και καταβάλουμε αυτή θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν υπάρχει πλήρης συμμετοχή και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θέλω λοιπόν να βασιστώ και στην δική σας την βοήθεια, προκειμένου το μήνυμα αυτό να περάσει ξεκάθαρα και στις δικές σας τις χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε πώς η πολιτική συνοχής μπορεί να συνδεθεί με το πρόγραμμα του Προέδρου Γιούνκερ. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της νέας αυτής πολιτικής έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο συνδέεται πλέον με την πολιτική συνοχής. Αποτελεί μόνο έναν πυλώνα βέβαια του όλου σχεδίου η πολιτική συνοχής. Το νέο πλαίσιο αυτό πολιτικής μας προσφέρει νέα μέσα, τα οποία δημιουργήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα έχουμε χρηματοδοτικά λοιπόν μέσα που θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια τη νέα αυτή επενδυτική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλε οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να χρησιμοποιήσουν τα νέα αυτά χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ε, μία νέα, θέλετε, διάσταση, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν τα δημόσια κονδύλια τα οποία δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, με κάθε ευρώ το οποίο επενδύουμε έχουμε όλο και μεγαλύτερη απόδοση. Με οποιαδήποτε μορφή και αν επενδύονται τα χρήματα αυτά, είτε στα πλαίσια ιδίου κεφαλαίων, είτε στα πλαίσια δανείων, τα νέα αυτά χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα σε όλους τους διαφορετικούς τομείς της περιφερειακής πολιτικής. Μεταφορές, υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενεργειακός τομέας και ούτε καθεξής. Ενδεχομένως η λειτουργία των μέσων αυτών να φαίνεται πολύπλοκη για κάποιες περιφερειακές αρχές, αλλά ήδη στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν ειδικευμένε ομάδες οι οποίες μπορούν τεχνικά να συνδράμουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τη μία χώρα στην άλλη, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη λεγόμενη μόχλευση. Ξέρω ότι Υπήρχαν ενησυχίε στην αρχή, ακόμα και εγώ ήδη είχα κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά τη λειτουργία αυτών των νέων χρηματοδοτικών μέσων. Πάντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν τα κράτη-μέλη, οι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα και θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλου του εταίρου, όλε τι εμπλεκόμενε αρχέ, προκειμένου να διαχειριστούν τα μέσα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυστυχώ στι 4 η ώρα θα πρέπει να αποχωρήσω, διότι έχω ένα γεύμα εργασία, μάλλον μια συνεδρίαση εργασία με τη νέα αυτή Task Force για την χρησιμοποίηση των νέων αυτών μέσων και θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, την τελευταία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική ευθύνη της επενδύσεις και τις, επενδύσεις και τις ε, δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε ότι τίθεται το θέμα της δημοσιονομικής ευθύνης και των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες χρειάζονται τη δική μας την υποστήριξη. Το θετικό νέο είναι ότι στα πλαίσια των κατευθυντήριων αυτών γραμμών και υποσκεκριμένων συνθήκων η εθνική συγχρηματοδότηση για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στον υπολογισμό του κρατικού δημοσίου ελλείμματος. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια νέα δέσμευση που είχε αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης οι χώρες που έχουν υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας διόρθωσης, διόρθωσης αυτού του δημοσίου ελλείμματος εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ στο όλο σχέδιο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και εσείς, το γεγονός των καθυστερούμενων πληρωμών. Δεν θα ήθελα να μου πείτε ότι δεν τον έφερα καθόλου το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι 90 δισεκατομμύρια ευρώ εκκρεμούν 19 δισεκατομμύρια ευρώ εκκρεμούσαν στο τέλος του 2014. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει αυτό το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει τα κονδύλια αυτά να απορροφηθούν. Σας ευχαριστώ πάντως για την συνεχή υποστήριξή σας στις πολύ δύσκολες Διαπραγματεύσει που είχαμε να κάνουμε για τον νέο προπολογισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να σταματήσουμε και το φαινόμενο αυτό των καθυστερούμενων πληρωμών και όλε τι αρνητικέ συνέπειες μπορεί να έχει σε άλλα προγράμματα. Χάρη λοιπόν στη δική σας την υποστήριξη καταφέραμε να σταματήσουμε το σημαντικότατο αυτό πρόβλημα και ήδη για το 2014-2020 για την περίοδο αυτή πρέπει να δεσμευθούν και τα τρία θεσμικά όργανα προκειμένου να μην προκύψει εκ νέου το πρόβλημα αυτό. Ήδη ανέλωσα αρκετό από τον χρόνο που μου είχατε δώσει αγαπητοί φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα, θέλει, θα ήθελα να έρχομαι συστηματικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τις νέες Open Days, τις νέες ημερίδες για τις ε, τον Οκτώβριο του 2015, όπως, είχαμε, όπως το είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Θα έχουμε βέβαια στο μέλλον τη δυνατότητα να αναλύσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις. Προσβλέπω σε έναν επικοδομητικό διάλογο μαζί σας για όλα αυτά τα ζητήματα που έθιξα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως να θέλετε να θίξετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με στη διάθεσή σας για ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, όπως ε, αναφέρατε ήδη εσείς, αλλά θα ήθελα και εγώ να το υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής. Θα πρέπει να φύγετε. Η Επίτροπος είναι πολύ απασχολημένη. Έχει άλλη σύσκεψη στην οποία θα πρέπει να παραστεί, πολύ σημαντική. Επομένως, θα έχουμε συζήτηση μαζί της για 45 λεπτά το ανώτερο. Ξεκινώ με τους ε, συντονιστές. Τους δίνω το λόγο για το πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ο κύριος Φανίλστερόι, παρακαλώ. Από πλευρά του ΕΛΚ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο που ήρθε εδώ και για ε, την ταχεία ε, έναρξη των εργασιών στο χαρτοφυλακείο της. Ε, σύντομα θέλω να κάποιες ερωτήσεις και ξέρω ότι και οι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Θα περιοριστώ εγώ. Για τις καθυστερούμενες πληρωμές σας πιστεύουμε ότι πάει στη σωστή κατεύθυνση και ότι εργάζεστε πολύ σκληρά. Μπορείτε όμως να μας παρουσιάσετε πώς έχει κατάσταση σήμερα. Σε ποιες χώρες δηλαδή γίνεται αυτό, ποιες χώρες ε, αφορά και πώς το διαχειρίζονται και πώς διαχειρίζεστε το υπόλοιπο. Γιατί όταν δεν έρχονται τα χρήματα και έχουν τελειώσει τα προγράμματα, είναι η κατάσταση δύσκολη. Σα έχω ξαναρωτήσει και μα υποσχεθήκατε ότι θα απαντήσετε. Μπορείτε σε 15 μέρε να μα φέρετε μια επισκόπηση τη κατάσταση, πώ έχει σήμερα και πώ έχει σε διάφορε χώρε. Γιατί ακούμε διάφορα μηνύματα ότι κάποιε χώρε θα βολεύουν μόνε του γιατί βάζουν δικά του λεφτά και κάποιε άλλε δυσκολεύονται. Εγώ θέλω πλήρη ενημέρωση εδώ στην Επιτροπή μα και επίσημη και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες μακροπεριφέρειες. Είναι γεγονός ότι είναι βασικό στοιχείο των πολιτικών μας αυτό, αλλά θέλω να κάνω την εξής σαφή δήλωση. Εμείς δεν θέλουμε η Ευρώπη να αποκτήσει ξαφνικά νέες μακροπεριφέρειες, ο καθένας ξαφνικά θέλει να ε, κάνει διασυνοριακή συνεργασία. Υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή και εργαλεία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι υπέρ της επέκτασης ε, αυτής της μακροπεριφέρεια. Και θα ήθελα και σε αυτό να δεσμευτείτε, να κάνετε μια δήλωση ξεκάθαρη. Παρακαλώ. Η Επίτροπος θα ήθελε να απαντήσει τώρα. Ίσως έχετε νέα στοιχεία να δώσετε στον κύριο ε, Νίστελ Ρόι. Θέλετε να απαντήσετε τώρα. Ναι, ή μήπω να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συντονιστές και απατάτες συνολικά στο τέλος. Η κυρία Φρέιλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχουν ε, εγκριθεί ήδη τόσα πολλά επιχειρησιακά προγράμματα. Η πρώτη μου ερώτηση. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου να μην τρέχουν τα ΕΣΠΑ ή να μην έχουν εγκριθεί, γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα με ενδιαφέρει αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα, στο μέλλον πώς θα ερμηνεύεται η ευελιξία στο σύμφωνο σταθερότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Ως κοινοβούλιο, ο Λάμπερτ Φανίστε και εγώ διαπραγματευθήκαμε το γενικό κανονισμό και προσπαθήσαμε να βρούμε και να εντάξουμε το λεγόμενο χρυσό κανόνα που πάνω κάτω έλεγε αυτό που ερμηνεύει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω όμως καταλάβει πάρα πολύ πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό χωρίς να προβάλλει κανείς καμιά αντίρρηση. Μπράβο σας, καταπληκτικό, γιατί αγωνιστήκαμε πάρα πολύ σκληρά, δεν το πετύχαμε στη διαπραγμάτευση, δεν πέρασε, αλλά θα με διέφερε τώρα πώς θα δημορφωθεί αυτό στην πράξη. Ευχαριστώ. και εκ μέρους ε, της πολιτικής ε, ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Ξέρετε, ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν βρει ακόμα την, ε, σωστή ταχύτητα, το σωστό ρυθμό στην απορρόφηση των κονδυλίων. Ενδεχομένω οι κυβερνήσεις τους δεν κάνουν τίποτα. Είναι ένα βάρο αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιο μέσο, κάποιο εργαλείο να εξαναγκάσει τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Μπορεί αυτό να γίνει μέσω της οικονομικής διακυβέρνησης. Από πλευράς άλλων, κύριος Νιούτον Μπόρκ. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε. Ελπίζω να σας βλέπουμε και συχνά τα επόμενα χρόνια. Καλή αρχή σημαίνει καλή συνεργασία. Ε, έχω την εξή ερώτηση. Το είπατε κι εσείς. Ε, είναι τραγική η αρχή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Έχουμε μείνει ένα χρόνο πίσω. Υπάρχουν κράτη που έχουν προβλήματα δυνατότητας απορρόφησης τι θα κάνετε τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν να επενδυθούν αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν. Δεύτερη ερώτηση. Ξέρω ότι μόλις αναλάβατε, αλλά σας λένε τι έχει γίνει στο παρελθόν και βγάζετε και τα διδάγματα από τις υπηρεσίες σας, σας ενημερώνουν. Τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα για να αποφύγουμε να τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Μετά από λίγα χρόνια, όταν θα προετοιμάζουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, να μην ε, ξαναδούμε αυτά τα πράγματα, να μην τα ξαναζήσουμε και όπως λένε και οι Γάλλοι, να μην επαναληφθεί αυτή η ιστορία. Άλλη ερώτηση. Πώς θα αποφύγετε, θα αποτρέψετε ε, στα κράτη-μέλη, γιατί είναι ανησυχητικά τα πρώτα μηνύματα, να μην γίνονται έλεγχοι επί ελέγχων. Ε, για την διαχείριση των κονδυλίων. Συχνά μιλάμε για ε, το διοικητικό και το γραφειοκρατικό άχθος. Αλλά όταν είσαι μικρομεσαία επιχείρηση, θες να ξέρεις, να έχεις ένα ε, προγραμματισμό και να ξέρεις ότι ισχύει και η αρχή της εμπιστοσύνης και όχι η έλεγχη επί ελέγχων. Δηλαδή όταν δηλώνει κάποιος κάτι, ε, σημαίνει ότι αυτό ισχύει καταρχήν και να μην είμαστε τόσο καχύποπτοι και τόσο δύσπιστοι. Και τι γίνεται με την ατζέντα για τις πόλεις και την πολιτική σας δέσμευση για ενίσχυση ουσιαστική της αστικής διάστασης ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτά τα ολίγα είχα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Σομάρτσε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ θερμά διότι ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Είχα διάφορες ερωτήσεις να σας θέσω για το χρονοδιάγραμμα. Εσείς έχετε ήδη απαντήσει. Θέλω να χαιρετήσω την προσπάθεια που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να επικυρώσει όσο δυνατόν περισσότερα προγράμματα μέχρι το τέλος του 2014. Υπάρχουν προγράμματα προς επικύρηση, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 220 δις θα πρέπει να γίνει ε, σωστή δουλειά για να μην έχουμε δυσάρεστες ε, εκπλήξεις όταν θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, είναι σημαντικό να έχουμε επιλογές επενδύσεων σωστές, τις οποίες να έχουν κάνει περιφέρειες στα διαφορά τους επιχειρησιακά προγράμματα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε προς ποιους στόχους κατευθύνονται τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Και η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το σχέδιο Juncker. Ξέρετε, οι ιδιώτες επενδυτές ενίοτε δεν θέλουν να αναλαμβάνουν μεγάλους κινδύνους και προτιμούν να διοχετεύουν τις επενδύσεις τους στις μεγάλες οικονομικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και στις μεγάλες περιφέρειες. Ενώ οι ανάγκες είναι εξαιρετικά σημαντικές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Επομένως ερωτώ, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κατευθύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε επικράτειες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ε, για παράδειγμα να ωφεληθούν και οι νέοι από αυτό. Μπορεί με την εγγύηση για τους νέους, με την εγγύηση για την νεολαία να ε, συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προεβλήματος. Όλοι παρακολουθήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην επικυρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι με την πολιτική συνοχή μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε οι νέοι από ε, μειονεκτούσες περιφέρειες ε, να ε, βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ και να μην προσελκύονται σε άλλες τάσεις και σε, άλλες, σε άλλα κινήματα. Και τέλος, τι ε, θα κάνετε για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάνα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε και από πλευρά μου στην, Επιτροπή μας. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις σας. Έχω μια πολύ ειδική ερώτηση για το επενδυτικό σχέδιο και για τον περιορισμό ε, και ε, τη διασύνδεση μάλλον με το Ταμείο Συνοχής. Πώς θέλετε να αποφύγετε μια διάλυση, ένα κατακαιρματισμό ή και παράλληλη ε, μορφή επενδυτικής πολιτικής που δεν θα είναι όπως η πολιτική συνοχής που διέπεται από κάποιους κανόνες. Παράδειγμα, εδώ στην Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια θελήσαμε να συνδέσουμε την πολιτική συνοχή με την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος, την αηφορία με τους στόχους 2020 και οργανωτικά ισχύουν και υπάρχουν ορισμένα βασικά κριτήρια όπως η αρχή της εταιρική σχέσης ή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας ε, και με πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης, άλλος στόχος ήταν η εδαφική συνοχή. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Στο νέο επενδυτικό τώρα πρόγραμμα που λανσάρεται και έχει δημιουργηθεί και ένα νέο ταμείο, ε, δεν υπάρχουν οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες. Και βλέπετε κι εσείς ένα κίνδυνο εκεί. Ε, μήπως υπάρξει παράλληλη ανάπτυξη δύο διαφορετικών ειδών επενδυτικής πολιτικής υπερβάλλω λίγο, ε, τα ε, ταμεία συνοχής και τα διορθωτικά για τα φτωχά κράτη-μέλη και το άλλο ταμείο το επενδυτικό για τα ε, πλούσια. Και αντί να έχουμε εδαφική συνοχή, έχουμε μάλλον εδαφική απομάκρυνση και απόκληση. Και όχι μόνο εδαφική, αλλά και κοινωνική ενδεχομένως. Ευχαριστώ, η κυρία Νταμάτο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ξέρετε ότι ε, εφόσον ήσασταν Ευρωβουλευτής ότι τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα για την Ιταλία. γιατί ξέρετε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εξάμεινη προεδρία της Ιταλίας. Δεν το λέω όμως γι' αυτό, αλλά τα προγράμματα αυτά αφορούν το σύνολο της Ευρώπης. Και πολλές φορές αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η ευθύνη φαίνεται να ρίχνεται περισσότερο στα ίδια τα κράτη-μέλη ή στις περιφέρειες όσον αφορά την χρήση των διαφόρων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όμως για την αγέννηση ορισμένων περιφερειών. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η βοήθεια το οποίο θα μπορούσε να δοθεί, και το είχαμε πει αυτό και την προηγούμενη φορά, για τα κράτη-μέλη εκείνα, για τις περιφέρειες εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση επαρκή στα ταμεία και θα ήθελαν να αυξήσουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι ερωτήσεις από πλευρά συντονιστών και πολιτικών ομάδων. Δίνω τώρα το λόγο στην Επίτροπο να, για να απαντήσετε, αν μπορείτε βεβαίως, να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ η Επίτροπος. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Το ψήφισμα του Νοεμβρίου είναι αυτό που μας παρακίνησε έτσι ώστε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα των καθυστερούμενων αποσβέσεων και όπως είπα και στην ε, παρέμβασή μου, στην ομιλία μου προηγουμένως, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις. είναι αντικείμενο σύσκεψης ε, μεταξύ εμού, μεταξύ της Επιτρόπου Γεωργίευα και των αρμοδίων διευθυντών των υπηρεσιών. χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε ε, την κατάσταση, να ε, υψώσουμε ένα εμπόδιο σε αυτή τη χιονοστιβάδα και έχουμε σαν νούμερο τα 19 δις. Μιλούμε δηλαδή για αιτήματα πληρωμών τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στα τέλη του 2014 για τους βασικούς τομείς πολιτικής γιατί δεν μιλάμε μόνο για την περιφερειακή πολιτική βεβαίως. Αυτό ήταν το νούμερο που μας ενδιαφέρει. Και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει το 2015 να καταρτήσουν ένα σχέδιο για να μειώσουν το επίπεδο των απλήρωτων λογαριασμών. Ε, σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 2007-2013. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως και να έχει το πράγμα. Σας διαβεβαιώ ότι Δεν έχω βέβαια τα νούμερα, τα συγκεκριμένα και τα αριθμητικά στοιχεία για τις επιδόσεις όλο, της κάθε χώρας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτι που επηρεάζει όλες τις χώρες και σας διαβεβαιώ ότι η υπηρεσία μου, η αρμόδια γενική διεύθυνση θα κάνει ό,τι μπορεί. Ο κύριος Νίλστερ Ρόι, μπορούμε να έχουμε τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία ε, τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Η Επίτροπος, ναι, Τώρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Είναι, η γνώμη μου είναι κάπως διαφορετική από τη σας και από άλλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι οπαδός της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες. Ε, ε, ξεκινήσαμε την μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιωνίων νήσων. Δυστυχώς, ήταν πολιτική απόφαση να μην υπάρξει διεύρυνση τα επόμενα πέντε χρόνια. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να έχουμε τα σωστά πλαίσια έτσι ώστε να εμπλέκουμε ε, τα κράτη-μέλη και μη. Ε, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω ρουμανικά. Ε, Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι τα κράτη που δεν αποτελούν μέρος, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις στρατηγικές για τις μακροπεριφέρειες έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν λύσεις και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Έχουμε τη στρατηγική για την Αδριατική και τις Ιόνιες νήσους. Τέσσερα, ε, μέλη, τέσσερα κράτη αποτελούν, ε, συγκροτούν αν θέλετε αυτή τη μάκρο περιφέρεια. Δύο είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιταλία και η Ελλάδα και μπορούν να, να βοηθήσουν ιδιαίτερα τις άλλες δύο χώρες. Είναι πολύ σημαντικό ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις μακροπεριφέρειες μπορούμε να φτάσουμε σε, σε ικανοποιητικές λύσεις. Έχουμε στρατηγική λοιπόν για το Δούναβι αλλά και τις ε, χώρες της Βαλτικής. Στο Μιλάνο είναι το αρχηγείο της ε, μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίων Νήσων και σύμφωνα με τις εντολές του Συμβουλίου πρέπει να προβλέψουμε μια μακροπεριφέρεια και αντίστοιχη στρατηγική για τις Άλπεις. Η περιφερειακή πολιτική είναι κάτι που είναι πολύ περισσότερο από τα χρήματα, αν θέλετε. Δεν είναι μόνο τα κονδύλια το θέμα. Σε πάρα πολλές χώρες δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν, να γίνουν αντικείμενο αξιοποίηση τα κονδύλια αυτά, γιατί οι αρχές δεν ήταν οι κατάλληλες. Δεν, είχαν, ε, δεν μπορούσαν να το φέρουν αυτό σε πέρας. Και τώρα σχετικά με το ερώτημα ε, της κυρίας Κρέλ, να σας πω ότι έχουμε κράτη-μέλη με χαμηλό ποσοστό εφαρμογής ε, της νομοθεσίας. Όντως η μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι η Task Force, την οποία συγκροτήσαμε στα τέλη Δεκεμβρίου, για να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν ε, έχουν ψηλό ποσοστό εφαρμογής ε, και απορρόφησης κονδυλίων. Ε, για τις χώρες που είναι μέχρι 60%. Και είπαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη-μέλη Είναι σημαντικό οι προσπάθειες να είναι κοινέ, να είναι από όλες τις μεριές να καταβάλλονται οι προσπάθειες. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε ούτε από τα κριτήρια ούτε από, από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μέσα σε ένα χρόνο, μάλιστα μέσα σε 11 μήνες, θα μπορεί κανείς να κάνει αυτό που δεν κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, στα 7 τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε τα πάντα, θα κάνουμε ε, ό,τι είναι δυνατό και ξεκινήσαμε με τις αποστολές εμπειρογνωμόνων, ε, ειδικών από την αρμόδια γενική διευθύνση, ε, μετέβηκα στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, και θα καταρτήσουν σχέδιο δράσης για κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε να απορροφήσει καλύτερα και γρηγορότερα τα κονδύλια. Ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση να αξιοποιήσει τη τεχνική βοήθεια και να αποστείλει προσωπικό ανθρώπινους πόρους σε αυτές τις 8 μονάδες ε, έτσι ώστε να ε, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων. Μίλησα λοιπόν για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, για τους απλήρωτους λογαριασμούς της πολιτικής συνοχής. Παρόλα αυτά, αυτό δεν επηρέασε αρνητικά την εκκίνηση, την έναρξη των νέων προγραμμάτων. Ε, προχωρούμε δηλαδή και στους δύο δρόμους. Ε, ε, ολοκληρώνουμε ε, τα, τις εκκρεμότητες για το πρόγραμμα 2007-2013 και ξεκινούμε ήδη το 2014-2020 και έχουμε μόνο απομονώσει όλα αυτά που έχουν καθυστερήσει για να τα δουλέψουμε. Τώρα, ως προς την ευελιξία έχουμε την πιο έξυπνη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό το υιοθετήσαμε στην τελευταία σύσκεψη του Σώματος των Επιτρόπων και ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Είναι σημαντικό ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αναγνωρίζουν τη σημασία της πολιτικής συνοχής και δίνουν ιδιαίτερο καθεστώς στην εθνική συγχρηματοδότηση. Δηλαδή στο κομμάτι της εθνικής χρηματοδότησης αυτό το κομμάτι έχει ιδιαίτερο καθεστώς θα απαλλαχθούν κάποια κράτη-μέλη από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Δηλαδή η εθνική συγχρηματοδότηση δεν θα προσμετράται ε, στο εθνικό έλλειμμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μου τέθηκε ένα ερώτημα για τα νέα κράτη-μέλη. Δύσκολο ερώτημα πρέπει να πω. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι βάρος. Κάποια όντως καθυστέρησαν να εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές, τα περισσότερα θα έλεγα. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο σκληροί. Έχουμε μία task force για τις ε, δικαστήριο εφαρμογή και πιστεύουμε ότι αυτή η task θα ευεργετήσει τα κράτη-μέλη, θα ε, τα βοηθήσει. Θα στείλουμε ομάδες από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, όπου η απορρόφηση των κονδυλίων είναι κάτω του 60%. έτσι ώστε να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης. Ναι, είναι ένα δίδαγμα αυτό που πρέπει να αντλήσουμε και αν συγκρίνουμε με την περίοδο 2007-2013 πρέπει να πούμε ότι έχουμε προόδους. Γιατί ε, γιατί το ποσοστό απορρόφησης στα επιχειρησιακά προγράμματα είναι 63% και για την ίδια περίοδο προγραμματισμού στο προηγούμενο στάδιο το ποσοστό ήταν 15%. Το λέω αυτό για να απαντήσω στο ερώτημα που έχει να κάνει με τα νέα κράτη-μέλη. Τέλος, για να απαντήσω ε, στο ερώτημα της Άλντε, των φιλελεύθερων, πώς θα μάθουμε το μάθημά μας, ποια διδάγματα θα αντλήσουμε και πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον για να αποφύγουμε καταστάσεις που θα ε, δημιουργήσουν προβλήματα. Σίγουρα θα υπάρχουν έλεγχοι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έλεγχοι θα υπάρχουν και θα γίνονται. Υπάρχουν και γίνονται για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη, οργανώνονται και άλλωστε οι περισσότερες παρατηρι... παρατυπίες που εντοπίστηκαν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν τα κράτη-μέλη είχαν δράσει πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διάφοροι τρόποι να οργανώσει κανείς έναν έλεγχο και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα ε, και να δει κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και υπάρχουν και πολιτικές πτυχές που ε, εμπλέκονται εκεί. Ε, πρέπει να δούμε αν ένα πρόγραμμα ε, συμμορφούνται με την νομοθεσία και αν ναι, εάν όντως είναι χρήσιμο και ηθικά σωστό να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα σε περίοδο κρίσης. Έχουμε ήδη κάνει αυτή τη συζήτηση, π.χ. Για, το χτίσιμο ε, εγκαταστάσεων γκολφ, για το άνοιγμα κομμωτηρίων ως ε, υποτίθεται επιχειρηματικότητα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, μας απασχόλησε αυτό. Κατά πόσο θα χρηματοδοτήσουμε ε, το χτίσιμο ε, εγκαταστάσεων γκολφ σε περιόδους κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ε, την ευθύνη να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και έχουμε και την εντολή του δικαστηρίου που μας λέει να μην χτίζουμε πλέον τοπικά αεροδρόμια, την Πολωνία, για παράδειγμα, δισεκατομμύρια επενδύσεων έχουν έχουν χρησιμοποιηθεί για να έχουμε 10-15 χιλιάδες επιβάτες την εβδομάδα μόνο. Όχι πια. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν μπορούμε πλέον να τις επιτρέψουμε. Δεν ξέρουμε τι επιθυμούν τα κράτη-μέλη να εντάξουν στην επικεφαλίδα καινοτομία και έρευνα. Σε κάθε περίπτωση το λέω ξεκάθαρα, δεν δεχόμαστε πλέον αυτό το οποίο παλαιότερα αποκαλούσαμε ε, αμφίβολες επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβει εκείνος τέτοιου είδους επενδύσεις και δεν θέλουμε αυτά να τα χρηματοδοτούμε με το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα ήδη κατά την παρουσίασή μου. Επιθυμούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να έχουν και να υποβάλουν ποιοτικά έργα ε, στην περίοδο 2014-2020, τα οποία και πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι διότι έχουμε την νομοθεσία ηλεκτρονικό τελωνίο ή ντουάν και μπορούν ε, τα κράτη-μέλη να ε, λειτουργήσουν πολύ ε, πιο αποτελεσματικά. Τώρα, ως προς τα επιχειρησιακά προγράμματα. Θέλουμε να μάθουμε και από τα κράτη-μέλη ποιες επενδύσεις σκοπεύουν να εξετάσουν και να έχουν για αυτή την περίοδο 2014-2020 και ε, μόλις μαθούμε στοιχεία, αμέσως θα τα διαβιβάζουμε και θα σας ενημερώνουμε στην Επιτροπή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες αυτές οι επενδύσεις ε, θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους 11 θεματικούς άξονες τους οποίους εγκρίνατε εσείς μαζί με το Συμβούλιο και εγγράψατε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στην επικεφαλίδα καινοτομία και έρευνα θα πρέπει να υπάρχουν μόνο πράγματα που να έχουν να κάνουν με καινοτομία και έρευνα και τίποτα άλλο. Σίγουρα η νεολαία είναι προτεραιότητα, οι νέοι είναι προτεραιότητα. Για την περιφερειακή πολιτική έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας με την Επίτροπο για τις κοινωνικές υποθέσεις για να έχουμε κοινά project με αποδέκτες τους νέους. Και ως προς τις μειονεκτικές περιφέρειες, τις μειονεκτούσες, αυτές που βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση. Ξέρετε ότι σε δύο εβδομάδες θα συμμετάσχω στη συνεδρίαση εκπροσώπων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί θα ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα τους προβλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτές τις περιφερειές. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο να ε, ε, στοχεύει αυτές τις εξόχως απόκεντρες ε, περιφέρειες. Τώρα, ως προς το επενδυτικό σχέδιο, το σχέδιο Juncker. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μηχανισμός αυτός καθεαυτός για να αξιοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Κάθε project, κάθε έργο πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά έτσι ώστε να δούμε εάν μπορούμε να κινητοποιήσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για το εν έργο. Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έρχεται να συμπληρώσει τα ήδη υπάρχοντα ταμεία για την περιφερειακή πολιτική και είναι σημαντικό ε, να ξέρουμε ότι δεν τα επηρεάζει. Έρχεται αφριστικά να συμβάλλει. Η κυρία Βάνα μου έθεσε ένα ερώτημα Να σας πω ότι αυτό που με ρωτήσατε δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή στην νομοθεσία. Υπάρχει στο σχέδιο Juncker, συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. για το πώς θα γίνουν όλα αυτά και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε οι επενδύσεις αυτές να μην οξύνουν τις διαφορές που ήδη υπάρχουν προσωπικά. Πιστεύω ότι πράγματι χρειαζόμαστε συζήτηση. Χρειαζόμαστε τις γεωγραφικές ποσοστώσεις. Έχουμε τον κανόνα του ε, όποιος ε, φτάνει πρώτος και σερβίρεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος, όμως αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Σίγουρα η νομοθεσία θα υιοθετηθεί μετά την ε, συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που σας ζητώ είναι να ε, μεριμνήσετε έτσι ώστε το αργότερο να είναι έτοιμο το νομοθετικό κείμενο σχετικά με το σχέδιο Juncker για να ξεκινήσουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι. Σίγουρα υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο το όπου, όπου θα ε, το οποίο θα δέχεται τα έργα, θα κάνει την επιλογή, θα δίνει τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη. Αυτό το γνωρίζετε ήδη, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ξέρουν ε, ότι θα πρέπει να στείλουν έργα σοβαρά, ε, με ένα φάκελο ε, σοβαρό και στέρεο για να μπορεί να είναι επιλέξιμος. Τώρα, ως προς το ερώτημα για την Ιταλία, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τρεις αυτές περιφέρειες, την Καλαβρία, την Σικελία και την Καμπανία. Θέλουμε να προβλέψουμε να οργανώσουμε μια ε, διάσκεψη, μια συνεδρίαση. Είναι οι περιφέρειες οι οποίες ε, ε, είναι οι τελευταίες που έχουν στείλει έργα για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Γιατί υπήρξε τέτοια μεγάλη καθυστέρηση, γιατί υπήρχε μπλοκάρισμα σε επίπεδο περιφερειακής διακυβέρνησης και μπλοκάρισμα σε επίπεδο συντονισμού με την εθνική κυβέρνηση, την κεντρική η συγχρηματοδότηση εθνική ήταν στο 50% την περίοδο 2007-2013, αλλά τα προγράμματα δεν απέδωσαν όσο ελπίζαν και έτσι το 5% της εθνικής ε, συγχρηματοδότησης μειώθηκε στο 25%. Το κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το ίδιο ε, σε τι ποσοστό θα συμβάλλει και θα συγχρηματοδοτήσει. Όμως ε, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό που θέλουμε είναι να βρεθεί λύση για αυτές τις περιφέρειες όπως έλεγα και στην ακρόασή μου, είμαι πεπισμένη ότι εμείς καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες. Δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε αυτές τις περιφέρειες στο, στη Νότια Ιταλία. Όμως δεν υπήρξε οικονομική ανάπτυξη περισσότερη, δεν υπήρξαν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Task Force πρέπει να αναλύσει, να το μελετήσει αυτό. Ε, ε, για αυτή την περιφέρεια την μεγάλη του Μετζοτζόρνο να μάθει γιατί ακριβώς συνέβη αυτό. Έχουμε άλλα παραδείγματα όπου έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε παραδείγματα όπου ε, οι ανισότητες μειώνονται κάθε φορά που γίνονται έργα στις περιοχές. Όταν τα κράτη-μέλη ε, δέχονται τεχνική βοήθεια, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Αυτή η κατάσταση λοιπόν στο νότο της ε, ε, Ιταλίας πρέπει να αναλυθεί περισσότερο για να δούμε πού είναι το κακό και να το κόψουμε από τη ρίζα του. Άλλες ερωτήσεις. Ε, προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις όλες φαντάζομαι. Ναι, προσπαθήσατε ε, να απαντήσετε σε όλες. Επιτρέψτε μου ένα μικρό γύρο ακόμα. ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Βαλκάρσελ και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, Βαλκάτσερτ, και ο κύριος Μπλάνκο Λόπες έχουν ερωτήσεις. Αν συμφωνείτε, να ακούσουμε και αυτούς τους τρεις, για να προλάβουμε να τελειώσουμε, παρακαλώ. Sí. Gracias, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την παρέμβασή σας αλλά και για την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει. Δεν θελήσατε να αποφύγετε κανένα θέμα όσο ακαθόδες και να ήταν και ήταν μερικά ακαθόδη. Και πραγματικά αξίζει να σας ε, ποτίσουμε τιμή και σεβασμό. Και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως στο έργο σας. Έχω μια ερώτηση και μια παρατήρηση. Την ερώτηση δεν θα την κάνω, γιατί με κάλυψε ο κύριος Βανίστεροι όταν αναφέρθηκε ε, στις καθυστερημένες ή κρεμούσες πληρωμές. Απαντήσατε όμως αυτό. Η ε, παρατήρηση. Κυρία παρατηρηση κυρια εμένα με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτό που είπατε για τις ε, open days, τις ανοιχτές ημερίδες των πόλεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, έχουμε αυτή ε, την ε, εκτίμηση προς την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι τώρα η 13η φορά που θα διοργανωθεί αυτή η ημεριδα 12 με 15 Οκτωβρίου με τίτλο ε, πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης εταίροι για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και χαίρομαι που και εσείς το αναφέρατε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέχεται σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι αυτές οι μερίδες ανοιχτών θυρών και ελπίζουμε να ξεπεράσουν τα 800 πρόσωπα ε, οι ε, επισκέπτες συμμετέχοντες. Ευχαριστώ κύριο Σπόλτσεκ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα τα πρότεινε το Δεκέμβριο και προβλέπει διπλασιασμό. Πώς το έχετε φανταστεί αυτό ακριβώς. Συγκεκριμένα εννοώ την εφαρμογή στην πράξη. Στα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί, πώς θα μεταφερθεί ε, ε, αυτό ο διπλασιασμός των κονδυλίων. Συγκεκριμένα μιλώ για έργα, για προγράμματα που τρέχουν. Και ελπίζω την επόμενη φορά να έχετε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν ερωτήσει και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όχι μόνο οι συντονιστέ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπλάνκολοπ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πληροφόρηση που μας ε, παρουσιάσατε για τις καθυστερημένες ε, κρεμούς πληρωμές. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι Κάτι που κληρονόμησε η Επίτροπος και δεν μπορούμε τώρα να απαιτούμε και πολύ σφοδρά μέσα σε δύο μήνες να λύσει αυτό που δεν μπόρεσε να λυθεί χρόνια τώρα. Οπότε οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ας μετριάσουν λίγο ε, τους τόνους. Λες και είναι νέο αυτό το πρόγραμμα και φταίει η σημερινή Επίτροπος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάντως για την ενημέρωση και θέλω να σας διαβιβάσω μια ανησυχία μου, στην οποία και εσείς αναφερθήκατε. Είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα σε χώρες που έχουν ανάγκη αυτές τις επενδύσεις ως αποτέλεσμα της υποαπορρόφησης στην προηγούμενη περίοδο ή την αντίστοιχη. Θα ήτανε πολύ αρνητικό να χάσουν αυτή την ευκαιρία, την επενδυτική που προσφέρει η πολιτική συνοχή. Ιδιαίτερα τη στιγμή που πολλέ από τις χώρες αυτές ε, είναι χώρε που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και μάλιστα περιέργως είναι χώρε του Νότου. Πώ προβλέπει η επίτροπο να βοηθήσει αυτέ τι χώρε, το θίξατε στην απάντησή σα, για να προλάβουν να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια πριν κλείσει οριστικά η προγραμματική αυτή περίοδος. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δέκα ακόμα συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε επρακή χρόνο. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη και σας υπόσχομαι ότι ήδη από αύριο θα αρχίσουμε να διοργανώνουμε τη νέα ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπό μας. Θα δούμε πότε το πρόγραμμά της μας επιτρέπει να διοργανώσουμε μια τέτοια ακόμα ανταλλαγή απόψεων. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την ε, Επίτροπο Κρέτσου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να την ξαναδούμε εδώ στην Επιτροπή μας πολύ σύντομα. Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε τώρα σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις ανοιχτές ημερίδες, τα Open Days που θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο, Πράγματι, πρόκειται για μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και με την Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Regio θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε σίγουρη επιτυχώς την εκδήλωση αυτή. Μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική για την οποία θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη πρόθεση είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής να τονίσουμε τη σημασία της περιφερειακής πολιτικής για τις περιφέρειες και για τους κατοίκους των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντική λοιπόν η εκδήλωση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που πολλά από τα νέα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζι επιθυμούν να εργαστούν για τη νέα αυτή εκδήλωση και έχουν ήδη μια πάρα πολύ καλή γνώση του τι απαιτείται προκειμένου η εκδήλωση αυτή να στεφθεί με επιτυχία. Πάντω, στην επαφή που θα έχω και με του εκπροσώπου τη Επιτροπή των Περιφερειών, βασικό μου μέλημα είναι να είμαι σε συνεχή επαφή με όσου εκπροσωπούν σε τοπικό επίπεδο τι περιφέρειε, δηλαδή και τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ, αλλά και του εκπροσώπου των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τι επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια συνδιάσκεψη στις Βρυξέλλες με όλους αυτούς εκπροσώπους που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοινού θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε τις ανοιχτές αυτές ημερίδες για τις πόλεις. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες ερωτήσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, επιθυμούσαμε όντως να διπλασιάσουμε τη συμβολή των μέσων αυτών στην περίοδο την οποία αναφέρεται όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα, πιο συγκεκριμένα, και όπως σας είπα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε δημιουργήσει πλέον μία πλατφόρμα προκειμένου να καταφέρουμε τεχνικά να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη. 420 εκπρόσωποι από τις μονάδες διαχείρισης όλων των κρατών μελών πρόκειται να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα αυτή και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουν άμεση επαφή με τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά τον τρόπο τα κράτη-μέλη και πιο συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές για την διαχείριση της ε, κοινοτικής χρηματοδότησης θα είναι σε θέση να έχουν πιο συχνές επαφές. Ξέρετε ότι όσον αφορά την αστική ανάπτυξη και όσον αφορά την ε, προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο στην προηγούμενη περίοδο ε, προγραμματισμού και μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέτρα όχι μόνο για αυτούς τους δύο τομείς, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο τομέα, ενέργεια, μεταφορές, αυτό όσον αφορά τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Ξέρω ότι αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέτρα είναι κάπως πολύπλοκα στην εφαρμογή τους, αλλά είμαι σίγουρη ότι τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να βρούνε ή να ανταλλάξουν μεταξύ τους τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Η Ισπανία, η Μάλτα και η Γαλλία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά και όντως φαίνεται στην πράξη ότι κάθε φορά που επενδύουμε ένα ευρώ η απόδοση είναι τρία ή τέσσερα ευρώ. Ο απότερος λοιπόν στόχος αυτών των νέων χρηματοτικών μέτρων είναι να λειτουργήσουν όπως σας είπα πολλαπλασιαστικά στα πλαίσια της πραγματικής οικονομίας. Και ξέρετε ότι έχουμε το Γιάσπερ, το Τζέσικα, το Τζέρεμι, όλα τα μέσα αυτά τα οποία κατά την άποψή μου δεν χρησιμοποιούνται ακόμα επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαν να υποφεληθούν ακόμα περισσότερο τα κράτη-μέλη από τα μέσα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα νέα αυτά μέσα, η απόδοση των επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα αποτελέσματα είναι θετικά και πολύ χειροπιαστά. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές που δεν έχουν καταβληθεί, όσον αφορά τα τιμολόγια τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί, Σίγουρα θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αυτό που έχουμε κληρονομήσει από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού Πάντως ξέρετε ότι δεν είναι απόλυτη δική μου αρμοδιότητα το μέσα αυτός. Νομίζω ότι σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη βοήθεια της κυρίας Γεωργίευα θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα διάλογο. Ήδη έχω έρθει σε επαφή μαζί της και έχουμε ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού να μας βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και νομίζω όμως ότι και η Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να συμβάλλει προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Θα έλεγα μάλιστα ότι το πρόβλημα αυτό θα έπρεπε να επιληθεί από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα το επενδυτικό σχέδιο Juncker, και εγώ προφανώς θέλω οι επενδύσεις να γίνουν κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται αυτή τη στιγμή να διδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία και να αρχίσει το πρόγραμμα αυτό και το σχετικό ταμείο να λειτουργούν ήδη από τον Ιούνιο. 315 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να δοθούν σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τα κονδύλια τα οποία ήδη υφίστανται στα πλαίσια προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί, που έχουν αρχίσει ακόμα να, που έχουν αρχίσει να τρέχουν ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αυτή ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη ενημέρωση. Μας υποσχεθήκατε να μας στείλετε πληροφορίες όσον αφορά τις καθυστερούμενες πληρωμές και όσον αφορά την γεωγραφική διάσταση των καθυστερούμενων αυτών πληρωμών μας είπατε σε δύο εβδομάδες, άρα περιμένουμε τις πληροφορίες αυτές και όπως σας είπα θα φροντίσουμε το στομότερο δυνατόν να διοργανώσουμε την επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Σας εύχομαι επιτυχή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε. Thanks.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Can we continue with the... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε με τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Thank you very much. Σας παρακαλώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι καθίστε προκειμένου να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Να δώσω όμως πρώτα το λόγο στον κύριο Βανίστερόη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα διαδικαστικό ζήτημα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθε προφανώς η Επίτροπος με όλες αυτές τις πολύτιμες και σημαντικές πληροφορίες. Αλλά όπως είπατε είχαμε ένα κατάλογο 10 ακόμα ομιλητών που ήθελαν να πάρουν το λόγο και είχαν προετοιμάσει και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είναι λίγο σαν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Είχαμε το πρώτο ημίχρονο αυτή τη στιγμή με την Επίτροπο. Θα θέλαμε όμως να περάσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο δυνατόν. Ενδεχομένως να μπορούσαμε δηλαδή να δώσουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους τη δυνατότητα να προωθήσουν και να υποβάλουν μάλλον τα ερωτήματά τους προς την Επίτροπο. Ξέρετε ότι είναι προβληματική κατάσταση για τους συναδέλφους εκείνους που είχαν προετοιμάσει συγκεκριμένε ερωτήσεις και δεν κατάφεραν τελικά να πάρουν το λόγο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση αυτή, αλλά σας το είπα ήδη, ότι ήδη από σήμερα θα ξεκινήσουμε να διοργανώνουμε την ε, δυνατότητα της επόμενης ε, συνάντησης που θα έχουμε με την Επίτροπο. Αυτό όμως εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα της Επιτρόπου και από το χρονοδιάγραμμα των δικών μας συνεδριάσεων. Πάντως, ε, προβλέπεται ήδη τους επόμενους μήνες να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο για συγκεκριμένα εξειδικευμένα ζητήματα. Θα διατηρήσω εγώ τον κατάλογο αυτό των συναδέλφων που δεν κατάφεραν σήμερα να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Μάλιστα θα μπορούσα να υποβάλω τα ερωτήματά σας γραπτός και να δούμε και τι απαντήσεις μπορεί να σας προωθήσει ενδεχομένως η Επίτροπος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την κατανόησή σας και ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίε κινητικότητα και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι θεμελιώδε δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πυλώνα της εσωτερική αγοράς. Η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται έκθεση για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης. Ο απότερος στόχος είναι να έχουν καλύτερη πρόσβαση εργαζόμενοι σε υπηρεσίες επαγγελματικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας Επιτροπή συντάσσει μία γνωμοδότηση και συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Νταντσίλα και ήδη τον Δεκέμβριο του 2014 μας είχε εκθέσει τις πρώτες, πρώτες της απόψεις και σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Προτείνουμε ερμηνεία κατάθεση τροπολογιών να είναι η, η 13η Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι Φεβρουαρίου μάλλον, 13 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε στα τέλη Φεβρουαρίου και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να εγκρίνει η Επιτροπή Απασχόληση στην έκθεσή τη, στη συνεδρίαση που θα έχει το Μάρτιο. 13 Ιανουαρίου, λέει η Πρόεδρος, 12 το μεσημέρι, είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Έχουμε 10 μέρες μπροστά μας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, το λόγο έχει η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Πρόεδρε, αλλά και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για την παρουσία τους. Ξέρετε, κάθε μέρα άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίοι διασχίζουν τα σύνορα για να εργαστούν στη γειτονική χώρα. 7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι το 2013 ζούσαν και δούλευαν σε άλλο κράτος μέλος από τη χώρα προέλευσής τους. Το 78% ήταν ενεργοί δραστήρια οικονομικά και το 60% είχαν ήδη μια θέση απασχόλησης. Όλα αυτά είναι εφικτά γιατί ε, τα μπορούν οι Ευρωπαίοι να ε, κινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν άδεια εργασία, χάρη στην ελευθερία της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2005 μέχρι σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα ε, μέλος. Μετά και κυρίως μετά από τη διεύρυνση του 2004 και το 2007. Ωστόσο, αυτή δεν είναι παρά μόνο το 3,7% του γενικότερου εργασιακού δυναμικού. Η ροή κινητικότητας μετά τις δύο διευρε... διευρύνσεις οδήγησαν στην ενίσχυση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 1% για την περίοδο 2004-2009. Σε πολλές περιφέρειες και σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε ότι απουσιάζει ε, εργασιακό δυναμικό με υψηλά προσόντα. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ενεργείας, αλλά και μεγάλος αριθμός θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί. 5 εκατομμύρια είναι οι νέοι άνεργοι. Και ο αριθμός των κενών θέσεων το μόνο που κάνει είναι να αυξάνεται από το 2009 μέχρι ε, σήμερα και κυρίως στις περιφερειές όπου η ανάπτυξη είναι ταχεία και όπου βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες, στην ε, ε, οικολογία, στην τεχνολογία και το καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους όσους αναζητούν θέσεις απασχόλησης. Ποιο είναι αυτό? Το EURES, το EVRES. Είναι η διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα. Είναι μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν εργασία. Είναι δωρεάν αν παρέχει πληροφορίες σε όλες τις χώρες σε 25 γλώσσες, φέρνει τους αναζητούντες εργασία σε επαφή με τους εργοδότες που ψάχνουν συγκεκριμένες δεξιότητες, καθοδηγεί τους αναζητούντες εργασία προς τομείς και επαγγέλματα όπου παρουσιάζεται έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και στηρίζει ε, το Γιούρες το έβρεση, τα προγράμματα κινητικότητας των νέων. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει 4 εκατομμύρια επισκέψεις ανά μήνα. Συμβάλλει σε 150.000 επαφές σε μηνιαία βάση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οδηγεί σε περισσότερες από 50.000 καλύψεις θέσεων εργασίας ετησίως, ενώ 750.000 βιογραφικά υποβάλλονται μηνιαίως στην διαδικτυακή πύλη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα τη μεταρρύθμιση του δικτύου Γιούρες, κάτι που θα αυξήσει τον αριθμό των εταίρων που θα παρέχουν υπηρεσίες κινητικότητας μέσω του Γιούρες και θα ενοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών απασχόλησης έτσι ώστε να καλυφθούν ε, ακόμα περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό αυτό επικυμαίνεται επί του παρόντο μεταξύ 30 και 40% του συνόλου των διαθεσίμων θέσεων. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί τη μεταξέλιξη του δικτύου Γιούρες και ε, ε, θέλει να εναρμονιστεί με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία. Όμως, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες τι σχέση θα έχουν με το συντονισμό, με τη δικτύωση, ποιος θα είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Όλα αυτά ακόμα είναι ασαφή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει τη συνεργασία με την Ισλανδία, την Νορβηγία και το Λίχτενστάιν που είναι εταίροι στο δίκτυο Γιούρες και την Ελβετία βεβαίως. με την πρόταση κανονισμού το Γιούρες θα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες, μεγαλύτερες δυνατότητες. Πιστεύω όμως ότι οι εθνικές και διασυνοριακές δομές πρέπει να έχουν επαρκές προσωπικό, αρκετούς πόρους για να αναπτύξουν αυτή τη νέα δραστηριότητα. Και πρέπει να έχουν και προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό. Έχω συζητήσει με τους εκπροσώπους των διαφόρων γραφείων γιούρες στα κράτη-μέλη. Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, Ίσως υπάρξει ανισορροπία ε, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συνοριακές αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες όμως έχουν και τις περισσότερες πληροφορίες για να τοποθετήσουν εργαζομένους στις διαθέσιμες θέσεις. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί σε έργα και σε προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση που έχει συσσωρευτεί για να βελτιώσουμε τη συνεργασία ε, με τους εταίρους σε άλλα κράτη-μέλη και για να μπορούμε να ε, υλοποιήσουμε νέα διασυνοριακά έργα. Αυτή η μεταρρύθμιση επιτρέπει πιο στενή συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται με την κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 40 ετών. Στόχος είναι να έχουν δεξιότητες, να έχουν προσόντα, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες με έξυπνο τρόπο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτού του δικτύου, τα οποία να είναι στη διάθεση όλων. Υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες, ξέρετε, που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και καλό θα ήταν αυτοί οι πολίτες να είναι ενήμεροι και μάλιστα ακόμα και στην Ήπεθρο να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του δικτύου. Η καλύτερη η καλύτερη διυπουργική συνεργασία θα διευκολύνει το δίκτυο ε, αυτό, θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν και εμποδίζουν βεβαίως εργαζομένους να ε, κινηθούν, να μετακινηθούν και να εργαστούν σε άλλη χώρα. Υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει έλλειψη έγκυρων στοιχείων και πληροφοριών. Δεν γνωρίζουν πολύ συχνά οι εργαζόμενοι πώς θα πληρώσουν τους φόρους, πώς θα ασφαλιστούν, ε, θα έχουν κοινωνική ασφάλιση στην άλλη χώρα. Όλα αυτά πρέπει να τα επιλύσουμε και πρέπει να τους διευκολύνουμε. Και δίνουμε ιδιαίτερη μέρημνα ε, στους νέους, οι οποίοι διατίθενται περισσότερο να κινηθούν και να μετακινηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύψεις θέσεων και για απασχόληση αλλά και για μαθητεία και για στάζ και για εξάσκηση και για άσκηση. Είναι μια εναλλακτική λύση αυτή για να μπορούν να βρουν θέση απασχόληση σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στο τέλος της μαθητείας είναι σημαντικό να υπάρχει πιστοποίηση. Το δίπλωμα αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπως γίνεται άλλωστε και με τις κλασικές μορφές εκπαίδευσης ήδη. Υπογραμμίζουμε ε, λοιπόν το γεγονός ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε τους νέους με αυτό το πρόγραμμα First Job Euros, το η πρώτη δουλειά μέσω του δικτύου αυτού. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, να διαδραματίσουν. Διασυνοριακές ε, σχέσεις και χαίρομαι διότι όλα αυτά αναγράφονται στο κείμενο του Συμβουλίου. Προτείνω ορισμό για τη ε, διασυνοριακή κάλυψη θέσεων, ε, προτείνω ορισμό για τη διασυνοριακή συνεργασία και για τις αρμόδιες αρχές. Σκοπός είναι να υπάρξει σωστή διαμεσολάβηση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς. Ε, να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτού του είδους η συνεργασία είναι κάτι που θα ωφελήσει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Γιατί θα ε, συμμετάσχουν διάφοροι εταίροι, κοινωνικοί φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να έχουμε και τα απαραίτητα οικονομικά. Ε, την απαραίτητη χρηματοδότηση. Μέσω των γραφείων συντονισμού ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβεβαιώσει ότι όλες οι δράσεις του Γιούρες θα χρηματοδοτηθούν αναλόγως με τους στόχους που έχουν τεθεί και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικού κεφαλαίου του προγράμματος EASY. και έτσι θα έχουμε τους ίδιους κανόνες παντού και θα αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα κονδύλια με τον ίδιο τρόπο προς όφελος όλων των εταίρων μας. Η σημερινή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υιοθέτηση του κανονισμού γιούρες, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες της απασχόλησης ε, του γιούρες. Ε, και να αυξηθεί η κινητικότητά τους. Η Λετωνική Προεδρία θέλει το αργότερο μέχρι το τέλος της θητείας της να έχει υιοθετηθεί αυτός ο κανονισμός Γιούρες και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το Συμβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει τη θέση του στις 11 Δεκεμβρίου 2014 στη σχετική σύσκευση. Το μόνο που μένει τώρα είναι να υιοθετήσει και το Κοινοβούλιο τη θέση του. Ε, και αυτή η απόσταση ε, στο χρονοδιάγραμμα οφείλεται στις εκλογές ε, της περασμένης χρονιάς. Αυτή η απόκληση δηλαδή. Πιστεύω όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να κομίσει προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη λεπτομερή παρουσίαση. Τρεις και έχουμε παρόντες. Είναι ο κύριος Χέτμαν, ο κύριος Όλι Ρεν και η Τέρι Ρέντκε. Uh, uh, uh, και εκπροσωπείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Άκερς από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης είναι μαζί μας. Δεν είναι. Παρευρίσκεται. Αρχίζουμε όμως από τους σκιώδεις ηγητές. Ο κύριος Χέτμαν. Εδώ είναι. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγητρία για την νομοδότησή της για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης. Πολύ ενδιαφέρουσες οι τροπολογίες που προτείνεται και προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικεντρώνεστε σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας και εταιρική σχέσης, διότι βλέπουμε ότι εξακολουθεί να αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που φεύγουν από τη χώρα τους για να εργαστούν σε κάποια γειτονική. Και επίσης ε, οι παραμεθόριες περιφέρειες είναι συχνά απομακρυσμένες από το κέντρο, μοιραία της χώρας και έχουν προβλήματα γενικότερα και προβλήματα στην αγορά εργασίας. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και πολλές δουλειές. Ας πούμε, συνεργασία με χώρες όπως είναι το Λιχτενστάιν και η Ελβετία μας ενδιαφέρουν πολύ. Θα κάνω και εγώ κάποιες τροπολογίες ε, για να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε πιο ευέλικτη τη διασυνοριακή αυτή συνεργασία. Επίσης, θέλω να είναι πιο ισόρροπη γενικά η γνωμοδότηση. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω είναι μια καλή βάση, μια αφετηρία για περαιτέρω συνεργασία και προσβλέπω σε γόνιμη συνεργασία με την εισηγητρία. Ευχαριστώ κυρία Ρέντκε, Θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει ως τώρα. Ήδη ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Γιούρες ως εργαλείο, ως μέσο για να φέρει πιο κοντά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που είναι απολύτως κρίσιμο για μένα. Τώρα, συζητήσεις είχαμε Ήδη από το Δεκέμβριο για το θέμα αυτό η ομάδα μου χαιρετίζει και καλωσορίζει ε, τις ε, προσπάθειες της συγγήτριας. Συμφωνούμε για τα βασικά ζητήματα. Μερικά μόνο που θα θέλαμε να διευκρινίσουμε και που έχουν για μας σημασία και χρειάζονται και περαιτέρω συζήτηση για την γεννητικότητα. Έγιναν πολλές μελέτες που έδειξαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ή ελλείμματα στην κινητικότητα είναι το γλωσσικό ζήτημα, η γλωσσομάθεια, όπως και το θέμα των διαφορετικών νόμων και κανονισμών. Το EURES στο μέλλον θα πρέπει να είναι μια πραγματική πλατφόρμα για να μπορεί ο κόσμος να βρίσκει κάποια άκρη σε αυτό το λαβύρινθο ε, των νομοθεσιών και των κανονισμών ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια περιφέρεια που μιλείται άλλη ε, γλώσσα από τη μητρική του εργαζομένου. Και μπορεί και χωράει η προσπάθεια συντονισμού στο Γιούρες. Ένα δεύτερο που θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό, τώρα που αρχίζουμε τις προσπάθειες για τον νέο κανονισμό, θα πρέπει να βεβαιωθούμε από την αρχή ότι υπάρχει σωστός μηχανισμός παρακολούθησης, έτσι ώστε σταδιακά να εντοπίζουμε ποια στοιχεία της νέας προσέγγισης είναι χρήσιμα και πώς βοηθούν τον κόσμο να αξιοποιήσει το δικαίωμα της ελευθερίας της κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πλατφόρμα μετά από αυτή την πρώτη αρχή. Ελπίζω στη συνέχεια της διαδικασίας και στη συζήτηση να έχουμε γόνιμες συζητήσεις. Ευχαριστώ για το πρώτο σχέδιο αυτό και την ανταλλαγή απόψεων και για όλη τη δουλειά που έκανατε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμασιτς από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Ideal... Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, σε έναν ιδανικό κόσμο οι νέοι θα μπορούσαν να πάνε εύκολα σε άλλα κράτη-μέλη προκειμένου να εργαστούν εκεί επειδή το θέλουν πραγματικά όχι επειδή αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Δυστυχώ όμω σε πάρα πολλέ χώρε δεν υπάρχουν πλέον θέσει απασχόληση για τους νέου. και επομένως προκειμένου να μην χαραμίσουν την παιδεία του οι νέοι αυτοί θα πρέπει πλέον να είναι πιο κινητικοί, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία απασχόληση του δίνεται στην Ευρώπη. Συμφωνούμε με την ιδέα αυτή, αλλά αντί να έχουμε μια προσέγγιση εκ των άνω, θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την επικουρικότητα και να μπορούμε επίσης να δούμε ποιες δυνατότητες μπορούν να δοθούν σε τοπικό επίπεδο, επίπεδο αυτό είναι δυνατό. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα με τον λεγόμενο τουρισμό κοινωνικής ασφάλισης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε προγράμματα που θα προωθήσουν την πραγματική έβριση απασχόλησης και όχι τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ψάχνουν να κάνουν άγραπη δωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μανίστερο ζήτησε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με μεγάλη χαρά Είδα, ε, ε, ε, εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας και στην Επιτροπή Απασχόλησης γίνονται μεγάλες προσπάθειες και από την ίδια την Επίτροπο να δώσει μια νέα ορμή. Θέλω πολύ συγκεκριμένα να παραπέμψω σε προγράμματα που έχουμε, όπως είναι το Interreg. Και η αγορά εργασίας και κατάρτιση είναι από τις βασικές προτεραιότητες στο Interreg. Πολύ ωραία τα λέτε σε πολλά σημεία της νομοδότησης για τα δύο συνοριακά, αλλά να αναφέρουμε και τα ίδια μας τα εργαλεία από την ίδια μας την Επιτροπή. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Όταν γίνεται λόγος για την κινητικότητα, δεν τρελαίνονται κιόλας, δεν ενθουσιάζονται τα κράτη-μέλη. Η συνεργασία τους δεν είναι ιδεώδης ούτε στο Γιούρες, ούτε στην εκτέλεση των ε, δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτό. Καμιά φορά πρέπει να τους τραβάμε και ταυτί και να τους πούμε δεν το κάνετε και περιτεραιότητα. Είναι θέμα εργασίας και βοηθάει και ενδιαφέρει και τους πολίτες και τη νέα γενιά που πιο εύκολα ε, ταξιδεύει και περνάει και σύνορα για να βρει δουλειά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και το Interreg αλλά και να, πώς να το να παρακινήσουμε, να τολμούμε να ε, αποτιμούμε και να αξιολογούμε και τις επιδόσεις των κρατών μελών. Ελπίζω ε, να σας φανούν χρήσιμα αυτά που λέω. Θα κάνω και τροπολογίες σχετικά. Ευχαριστώ κύριο Τσέλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευγνωμονώ που ο συντονιστής μου ο Λάμπερτ Βαλίνστερ Ρόιτ αναφέρθηκε στα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και απόφασισαμε εμείς. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και την Ευγνωμονό που αναφέρθηκε στην διασυνοριακή συνεργασία και εστίασε τόσο πολύ και το θεωρεί τόσο κομβικό αυτό το θέμα. Γιατί κανονικά αυτό είναι το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εργαζόμαστε πέρα από σύνορα. Και αν ε, δούμε τι γίνεται με την επικουρικότητα, και εκεί υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κανονισμό που έχει να κάνει με την εδαφική συνοχή και ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές και ε, που θα πρέπει να διευκολύνει ε, τη συνεργασία. Είναι ο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την Περιφερειακή Συνεργασία. Για πρώτη φορά και την εδαφική συνεργασία έχουν ε, τη νομική δυνατότητα οι περιφέρειες και οι παραμεθόριες να υπάρχει νομική κάλυψη για τη δημιουργία και εταιριών ε, και ε, επιχειρήσεων για να αναλάβουν συγκεκριμένα έργα. Επειδή μόνο εισηγητή γνωρίζω πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον ε, των περιφερειών να το κάνουν αλλά και πόσο μεγάλες είναι οι αντιστάσεις και τα εμπόδια των κεντρικών κυβερνήσεων που δεν θέλουν να αφήσουν τις περιφέρειες να δράσουν αυτόνομα. Εμείς που είμαστε όμως περιφερειακή επιτροπή θα πρέπει να το εντάξουμε στις εργασίες μας και να μας απασχολήσει αυτό. Γιατί συχνά όταν δύο παραμεθόριες περιφέρειες θέλουν να διαχειριστούν θέματα υγείας, αποβλήτων, από κοινού ή μεταφορών και συγκοινωνιών, ε, πολύ συχνά είναι διαφορετικά τα εθνικά νομικά συστήματα. Και βεβαίως επιμένει κάθε κράτος να ε, κυριαρχήσει και να εφαρμοστεί ο δικός του νόμος. Αυτό είναι εμπόδιο για τις περιφέρειες. Μπορούν οι περιφέρειες πλέον να αποφασίζουν μόνες τους ε, ποια νομική βάση θέλουν, ε, με βάση ποια νομοθεσία και να προχωρήσουν σε μια κοινή προσπάθεια. Όπου γίνεται αυτό και είναι απαραίτητο θα πρέπει να το τονίζουμε και επίσης όταν πρόκειται για την κινητικότητα των εργαζομένων, τη διευκόλυνση της απασχόλησης, θα πρέπει και αυτό το μέσο που έχουμε να το αναφέρουμε. Προσωπικά θα το πράξω. Αυτό θα κάνω τροπολογίες στην κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Τσέλε υπάρχει μια ένταση μεταξύ των κεντρικών κυβερνήσεων, των πρωτεύουσών δηλαδή και των παραμεθόριων περιοχών. Και μια που έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ παρόντα, θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για την εστίαση και την προσέγγιση γιούρες. Είναι πολύ καλή έκθεση της συναδέλφου, δεν λέω, δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την πρότασή σας, με βάση το EURES θα μπορέσουν να καλυφθούν 30 με 40% των θέσεων εργασίας που παραμένουν κενές. Ε, δεν είδα πουθενά όμως συγκεκριμένο στόχο και ποσοστό ή ε, αριθμό. Έχετε καμιά ιδέα ε, σχετικά με αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα ερώτημα το οποίο έχω σε σχέση με την καταπληκτική αυτή γνωμοδότηση της κυρίας Νταντσίλα που προτείνει και πάρα πολλές τροπολογίες. Ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι μετά το δημοψήφισμα που έγινε στην Ελβετία για την κινητικότητα των εργαζομένων, η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί στη χώρα αυτή σε σχέση με την κατάσταση που ισχύει στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως λοιπόν στις τροπολογίες που καταθέτουμε, τουλάχιστον κάπου θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αναδιοργάνωση της σχετικής αυτής υπηρεσίας Γιούρες όταν συνεργάζεται και η Ελβετία με το πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα να δεσμευτεί η Ελβετία παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματός να εφαρμόσει τη Συμφωνία Γιούρες στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κινητικότητα των νέων αλλά και γενικότερα την κινητικότητα των εργαζομένων. Πίσω λοιπόν θα καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και το ζήτημα αυτό στις ε, τροπολογίες ε, τις οποίες θα καταθέσουμε για την έκθεση αυτή. Δεύτερον, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα ενδεχόμενης ε, σύγκρουσης μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Επομένως θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μια τυπική, αν θέλετε, περιφερειακή αρμοδιότητα, διότι οι περισσότεροι παράγοντες εδώ πέρα δραστηριοποιούνται σε ένα περιορισμένο εδαφικό τομέα. Πολλές φορές, ναι, διασυνοριακά, αλλά και πάλι σε ένα πολύ σαφές οριοθετημένο πλαίσιο. Συνεπώς, θα πρέπει να πούμε ότι ε, οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να διοργανώσουν διασυνοριακές υπηρεσίες για την απασχόληση στα πλαίσια του προγράμματος αυτού του Γιούρης. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος. Contribute to the discussion. Άλλος συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο. Thank you. Uh, Ms. Ευχαριστώ, εισηγήτρια. Θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις. To the comments. Ή στα σχόλια. Ευχαριστώ. Στις συζητήσεις που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της Ελβετίας, ε, έμαθα ότι θα υπάρξει μια νέα συμφωνία, όπως και με την Νορβηγία. 200.000 είναι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που ε, περνούν τα ελβετικά σύνορα από τη Γαλλία και τη Γερμανία και εργάζονται στην Ελβενία. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η συμφωνία με τη χώρα αυτή. Ελπίζω η συμφωνία να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό, αλλά και ότι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούν να μας ενημερώσουν ε, και να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας και ελπίζω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αναζητούντων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου είναι η τελευταία μέρα η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και αν ε, το κάνουμε αυτό μπορούμε να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Φεβρουάριο και θα είμαστε ε, εντός του χρονοδιαγράμματος. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή. Προχωρούμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, η συνάντηση των συντονιστών, η οποία θα λάβει χώρα και κλεισμένων των θυρών. Νωρί σήμερα ολοκληρώσαμε τις εργασίες της Επιτροπής. Καλό λοιπόν τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα.